προχωρούμε. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. Yeah, yeah,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 Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Έχουμε ψηφοφορία. Σας παρακαλώ να ελέγξουμε αν λειτουργεί το σύστημα. Τοποθετήστε τις κάρτες σας στη συσκευή, παρακαλώ. The is open, right, so Δοκιμαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Yeah, it works. Λειτουργεί το σύστημα και δεν ε, βλέπουμε να υπάρχει καμία κατάχρηση από πλευρά ε, κάποια πολιτική ομάδα υπό τη μορφή υπερβολικά πολλών ψήφων. Ξεκινάμε λοιπόν από τη θέσπιση μηχανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβιβασμό συμβαστική α. Σε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. 10 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ελέγχουμε την τροπολογία 10. And it is adopted. Εγκρίνεται. Ενρίκε, νόμιζα ότι μόνο εσύ ήσουν υπέρ. Αλλά βλέπω ότι πολλοί σε υποστηρίζουν. Τροπολογία 11, υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε πάλι, δεν είναι σαφές. Τροπολογία 11. Αρχή της ψηφοφορίας. close the Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια πλειοψηφία, εγκρίνεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. 13. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. 10 υπέρ, 9 κατά δεν ήταν τόσο προφανές. Ε, συμβαστική Β υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Το δεύτερο τμήμα της 18 υπέρ. Διότι το πρώτο καλύπτεται από την συμβαστική Β. Υπέρ λοιπόν της 18. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική γάμα, σι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D, δέλτα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 38, στην επόμενη σελίδα, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 39, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 40, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 41 παρακαλώ αρχή της ψηφοφορίας λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβαστική ή e, ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 47 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 9 υπέρ 9 κατά. Συμβιβαστική F υπέρ. Κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα της F υπέρ. F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης. Να ελέγξουμε επαλήθευση. Δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής τροπολογίας F. Λήξη της ψηφοφορίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία σύγχυση, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Προχωράμε λοιπόν στην 51. Δεύτερο τμήμα της 51, υπέρ. Κατά. Αποχές. Πράσινη. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Πάλι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται σαφώς. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η, όχι 63 υπέρ κατά απορρίπτεται νομίζω 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Επαλήθευση της 72 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 10 υπέρ, 8 κατά. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Επαλήθευση της 78 αρχή της ψηφοφορίας. Two people not voting. Δύο δεν έχουν ψηφίσει. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 9 υπέρ 10 κατά. 80 ε, υπέρ. Επαλήθευση της 80. Πάλι είναι πολύ μικρή διαφορά. Εγκρίνεται 10 υπέρ 9 κατά. 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και η τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε έναρξη της ψηφοφορίας. Όχι. Με τι να σας πω, με αυτή τη γραμματεία είμαι υποχρεωμένη να συνεργάζομαι. people don't vote. Oh, Τα δύο τρίτα έχουν ψηφίσει μόνο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της γνωμοδότησης. work here. Δεν λειτουργεί. Πρέπει να πατήσετε το κουμπί. Which one? Yeah, now everybody Yeah. Ωραία, ψήφισαν όλοι οι παρόντες. Λήξη της ψηφοφορίας λοιπόν. 13 υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές. Και μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. Έλεγχο τη εφαρμογή του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αίτηση έκθεση για το 2014. Συμβαστική Α. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Επειδή είναι συμβαστική, θα ήθελα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Νόμιζα ότι ήταν σαφές, αλλά αν ήταν μικρή τροπολογία θα το άφηνα, αλλά απορρίπτεται 7 υπέρ, 12 κατά. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα όλες τις ψηφοφορίες. Σε τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2, ε, η τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. 3 υπέρ. 3. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση της 3. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση της 8. Αρχή της ψηφοφορίας, λήξη, εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ. Κατά επαλήθευση της 13. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 9 υπέρ, 10 κατά. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά πίπτη 15 επειδή υιοθετήσαμε τη 14. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά επαλήθευση του δεύτερου μέρους της τροπολογίας 17 υπέρ. Ε, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση επίσης. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο πριν ε, ψηφίσουμε. Ε, αποφάση η πολιτική μας ομάδα να καταψηφίσει αυτή την ε, γνωμοδότηση και είναι ξεκάθαρη θέση της ομάδας μας. Είπαμε να καταψηφίσουμε κάθε γνωμοδότησε κάθε έκθεση, κάθε κείμενο από την πολιτική ομάδα της κυρίας Λεβεντέμου και το ξαναλέμε. Αυτή είναι η στάση μας επομένως και στην Συνταγματική Επιτροπή εναντί της ε, άκρας δεξιάς. Ευχαριστούμε. Άνεμας. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα την ε, Γραμματεία για την συνεργασία την οποία είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες και τι, τι, τι ψάχνετε το, την αγγλική μετάφραση ε, σε τι γλώσσα να σας τα πω πειράζει να σας τα πω στα Ολλανδικά όχι, α, ωραία δεν ξέρω πως είναι τον κύριο Πρέντε να τα πω στη γλώσσα μου ωραία, θα τα πω στα Ολλανδικά Οπότε σας έλεγα τη συνεργασία με την γραμματεία την ε, περασμένη εβδομάδα και τις ευχαριστίες μου πάντως. Θα ήθελα να σας επισημάνω το εξής. Είπαμε για συμβαστική τροπολογία. Πάντως δεν υπάρχει κάποιο πίμαχο σημείο θεωρώ μέσα στο κείμενο. Και άκουσα τον κύριο Πρέντα. Τον είδα πώς αντέδρασε. Νομίζω ότι η πολιτική μας ομάδα θα λάβει υπόψη αυτά το είπε ο κύριος Πρέντα για το πώς θα το βοηθούμε εμείς στο Κοινοβούλιο. Άκουσα με προσοχή και στην Συνταγματική Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα με αυτή τη γνωμοδότηση. Δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, να χρησιμοποιούμε κανόνια, να σκοτώσουμε μια μύδα. Και προετοιμάσαμε αυτή την ε, έκθεση με μια φυσιολογική διαδικασία. Οπότε τι να σας πω, αυτά τα οποία είπατε εσείς, εγώ δεν τα εισέπραξα. Σας ε, διαβεβαιώνω ότι και αυτό το οποίο λέτε εσείς, τα ξέρω τι γίνεται με τους λαϊκιστές. Ξέρετε, επί τρία χρόνια ζω με αστυνομική προστασία Ακριβώ γιατί με έχουν απειλήσει λαϊκιστές. Επομένω αυτά να μην τα λέτε σε μένα. Επομένως δεν υπάρχει θέμα και πρόβλημα ούτε στην ουσία του επί του τύπου. Ε, κύριε Κάφμαν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ πριν από την τελική ψηφοφορία εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδος να πω ότι και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει κανείς να κυνηγάει τα σπουργίτια με τα κανόνια. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια αντιπαράθεση σε μια πολιτική ομάδα η οποία προβάλλει ρατσιστικά συνθέματα και ως σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες θα τα πολεμήσουμε πάντοτε αυτά. Κάτι που παίζει ένα σημαντικό ρόλο εδώ για την Επιτροπή Συνταγματικών. Έχουμε απέναντί μας μια πολιτική ομάδα η οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να καταστρέψει, τα έχει πει αυτά η ίδια η κυρία Λεπέν, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε φιλοευρωπαίοι, θέλουμε να διατηρηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό με την παρούσα ψηφοφορία θέλουμε να δώσουμε ένα καθαρό μήνυμα υπέρ τη Ευρώπης. Listen, the idea of elected people are that fund... Η, ιδέα των δημοκρατικά εκλεγμένων είναι ότι διαφωνούμε θεμελιωδώς και ε, και εγώ διαφωνώ με άλλες πολιτικές ομάδες, αλλά εάν αρχίσουμε να αντιδράμε έτσι στους εισηγητές, τότε υπάρχουν πολλοί με τους οποίους ε, δεν θα ήθελα να συνεργαστώ στο Κοινοβούλιο, όχι μόνο στην ομάδα ΙΕΝΕΦ, αλλά και σε άλλες ομάδες. Και θα πρέπει να πω ότι οι παρατηρήσεις αυτές Τώρα, μετά από εβδομάδες εργασίας της Επιτροπής πάνω στην έκθεση αυτή, είναι πεδαριώδες. Έχουμε συντονιστεί από την ομάδα S&D, από την ομάδα ΕΛΚ, που στην ε, συνάντηση των ε, συντονιστών συμφώνησαν ότι ο κύριος Άνεμανς μπορεί να είναι εισηγητής ε, της έκθεσης αυτής. Γιατί δεν μας είπαν τότε ότι η συνέπεια της απόφασης αυτής θα ήταν ότι θα καταψηφίσουν. Το θέμα δεν είναι ο Άνεμανς, ούτε η ΕΛΚ, ούτε το SND Είναι το θέμα ότι η ε, Επιτροπή ΑΦΚΟ ε, φέρεται με τρόπο πεδαριώδη και ε, και ρεζιλευτικό για το σύνολο του Κοινοβουλίου. Δεν θα ξεκινήσω τώρα εις βάθος ε, ιδεολογική συζήτηση. Οι πράσινοι θα καταψηφίσουν ε, την, ε, την αυτή επειδή καταψηφίστηκε η τροπολογία 16 δική μας. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη από την ΚΟΕ. Εγώ ήθελα να σας πω ότι και εγώ θα καταψηφίσω και στην ε, Ολομέλεια. Θα ψηφίσω και τις τροπολογίες του Εθνικού Μετώπου. Οι συμβαστικές τροπολογίες δεν μου φαίνονται τόσο εύστοχες. Από την άλλη μεριά, βέβαια, δεν συμφωνώ με το ότι θα πρέπει να ψηφίζουμε ναι, όχι ανάλογα με το ποιο ε, έχει συντάξει ένα κείμενο. Προσωπικά θα καταψηφίσω γιατί πολλές δικές μας τροπολογίες ε, και κυρίως ε, του Τέρι Κάμπρας δεν έγιναν αποδεκτές. Δεν θέλει άλλο το λόγο, τότε θα ψηφίσουμε τελική ψηφοφορία γίνεται τώρα και θα γίνει ηλεκτρονικά. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. So it's, it's rejected by 15 to... Απορρίπτεται. 15-4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 Αυτή ήταν η τελευταία ψηφοφορία. Ναι. Λέει ο γραμματέας προχωράμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Ah, Παρακαλώ, θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως ε, την συνάντηση των συντονιστών, διότι... Πρέπει να είναι σύντομη η συνεδρίαση αυτή. Πρέπει να πάμε μετά στη συνάντηση για την Ουκρανία. Έναρξη της συνεδρίασης των συντονιστών. Παρακαλώ, όποιος δεν είναι συντονιστής, να αποχωρήσει. To do something to make them, uh, to teach them how to behave, so that they have to respect the rights of member state, of member of parliament.